Αγαπητοί συνάδελφοι, ο πρόεδρος μου ζήτησε να κάνω την ακόλουθη δήλωση. Αγαπητοί συνάδελφοι, η ερχόμενη Κυριακή είναι η Διεθνής ημέρα κατά της βίας εις βάρος των γυναικών. Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα όμως αυτή η βία στον κόσμο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γνωρίζει κοινωνικά και πολιτισμικά όρια. Εκτιμάται πως μία στις πέντε γυναίκες μία φορά στη ζωή της έχει πέσει θύμα βίας. Μιλάμε δηλαδή για σωματική ή ψυχολογική βία ή σεξουαλική παρενόχληση. Θα ήθελα τώρα να σας αναφέρω το άρθρο 1 της Χάρτας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αναφέρει πως είναι απαραβίαστη η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Άρθρο 3 ε, κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα στην ε, προσωπική του αυτοτέλεια και στην σωματική και ψυχική ακαιρεότητα. Έχουμε κάνει πολλά, αλλά πρέπει να κάνουμε ακόμη περισσότερα και βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει τέλος σε αυτή την βία. Θα πρέπει λοιπόν μαζί να παλέψουμε άνδρες και γυναίκες. Πρέπει λοιπόν να εφαρμόσουμε τα απαραίτητα μέτρα όλοι μαζί, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, κράτη, μέλη και κοινωνία των πολιτών να αναπτύξουν μια κοινή στρατηγική. Αυτή ήταν η δήλωση. Κύριε Γκουλάρ, επί της διαδικασίας. Κύριε Πρόεδρε, εγώ βρίσκω πάρα πολύ διασκεδαστικό το να κάνουμε δηλώσεις που αφορούν τη βία κατά των γυναικών τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε ότι δεν θα υπάρξει καμία γυναίκα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ε, Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αγκουλάρτ. Σας ζητώ ε, να, να ζητάτε το λόγο για διαδικαστικό όταν πράγματι πρόκειται για διαδικαστικό και να δείξετε την απαραίτητη αυτοπιθαρχία. Θέλω να χαιρετήσω και μια αντιπροσωπεία από την Ελβετική Ομοσπονδία που βρίσκεται στα θεωρία και χαιρετίζω τον πρόεδρο του Ελβετικού Εθνικού Συμβουλίου. και τους άλλους βουλευτές οι οποίοι είναι παρόντες από το Ελβετικό Εθνικό Συμβούλιο.